Στην την Τρίτη σύμφωνα με το άρθρο 54 θα υπογράψουμε πέντε πράξεις νομικές και στα πρακτικά μπορείτε να βρείτε και όλες ε, τις ε, λεπτομέρειες καθώς και τους τίτλους αυτών των νομικών